επίπτωση της μεταναστευτικής κρίσης στον τομέα των μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλό λοιπόν την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να πάρει το λόγο. Παρακαλώ κύριε Επίτροπε. Έχετε το λόγο. Κύριε Τάισεν. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, χαίρομαι για αυτή την ευκαιρία που μου δίνετε να συζητήσω μαζί σα για την επίπτωση τη μεταναστευτική κρίση στον τομέα των μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπω όλοι γνωρίζετε, δεδομένη τη δίχω προηγουμένου ροή μεταναστευτική, οι χώρε μέλη, κάποιε, έχουν επαναφέρει ελέγχου, ορισμένε προσωρινά και έτσι δυσκολεύεται η λειτουργία του χώρου Σέγγεν. Οι απειλές στην ασφάλειά μας οδήγησαν λοιπόν σε περιορισμό κάποιων μέσων μεταφοράς. Η... Ο τομέας της μεταφοράς είναι πολύ ευαίσθητος σε αυτό το θέμα. Οπότε η επανασυγωγή ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα γενικευμένα και σε πιο μόνιμη βάση καταλαβαίνετε ότι θα εμποδίσει και την κινητικότητα των Ευρωπαίων πολιτών αλλά θα δυσκολέψει και πάρα πολύ την ελεύθερη ανταλλαγή αγαθών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάνω από 2-3, 800 δισεκατομμύρια αξίας αγαθών και 700 εκατομμύρια τόνοι αγαθών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν έχει εκτιμήσει τη ζημιά από την επανεισαγωγή τέτοιων ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα και από ό,τι φαίνεται υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις στα σύνορα που επηρεάζουν και τις ε, μεταφορές ε, και τα μέσα μεταφοράς αλλά και τους ίδιους βέβαια τους επιβάτες. Και αυτό πλήττει πολύ σοβαρά την οικονομία μας. Έλεγχοι στα σύνορα επίσης απαιτούν παραπάνω χρήματα από τον προπολογισμό των κρατών μελών για να υπάρξουν οι κατάλληλες υποδομές και να πληρωθεί το ανθρώπινο δυναμικό. Έπειτα τα αγαθά δεν φτάνουν στην ώρα του, στον προορισμό τους, κάτι το οποίο πλήττει την ανταγωνιστικότητά μας. Και τέλος, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν τη σπονδυλική στήλη των μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση πλήττονται περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Έχουν πολύ μικρά περιθώρια κέρδους, οπότε κάθε αύξηση δαπανών έχει επιπτώσεις και στον τελικό καταναλωτή, αλλά και στην ίδια την ύπαρξη των ε, επιχειρήσεων μεταφορών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμάει ότι εφόσον υπάρξουν πλήρως έλεγχοι για να ελεγχθεί η μετακίνηση του κόσμου εντός του χώρου Σέγγεν, αυτό θα είχε μεγάλες επιπτώσεις στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης της τάξης 5 με 18 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Μακροπρόθεσμα βέβαια είναι πιο δύσκολο να εκτιμήσουμε το κόστος. Αλλά από τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα έχουμε καταλήξει στο ότι πόσο να επαναφερθούν οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα οι αρνητικές επιπτώσεις θα πλήξουν συνολικά την Ευρωπαϊκή Ένωση και την οικονομία της. Οι εμπορικές συναλλαγές θα μειωθούν, το κόστος θα αυξηθεί και κυρίως θα επηρεαστούν οι χώρες μέλη οι οποίες εξαρτώνται κατά πολύ από τις εσωτερικές μεταφορές. 1,7 δισεκατομμύρια πολίτες που δουλεύουν διασυνοριακά θα πληγούν από τέτοια μέτρα, κυρίως από χώρες όπως είναι η Σλοβακία, η Ουγγαρία, το Βέλγιο αλλά και άλλες όπου πολύ συχνά οι κάτοικοι δουλεύουν στις συνοριακές χώρες. Το εμπόριο επίσης θα πληγεί από τέτοιους ελέγχους. Συνεπώς, αυτές οι πρώτες εκτιμήσεις μας δείχνουν πόσο σοβαρά αρνητικές θα ήταν οι επιπτώσεις από την άρση της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός του χώρου Σέγγεν κάτι που είναι πολύ βασικό ως στοιχείο για την οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα για τις επιδόσεις του τομέα μεταφορών. Γι' αυτό λοιπόν, αν κλείσουν τα σύνορα μεταξύ χωρών μελών, αυτό πρέπει να είναι το πολύ μεταβατικό μέτρο, προσωρινό και να σταματήσει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν επ' αυτού στην ανακοίνωσή της της 4ης Μαρτίου και στο χάρτη πορείας για την επιστροφή στο Σέγγεν έχει επιμείνει στο ότι πρέπει να επιστρέψουμε πριν τα τέλη του 2016 στην κανονική κατάσταση με την πλήρη λειτουργία του χώρου Σέγγεν. Όσο διατηρούνται οι έλεγχοι, τόσο πιο δύσκολο και τόσο πιο πολύ θα μας κοστίσει η επαναφορά στον ε, ελεύθερο χώρο Σέγγεν. Οι οικονομικοί εταίροι όσο προσαρμόζονται στη νέα κατάσταση, ε, τόσο περισσότερο δύσκολο θα τους είναι να επιστρέψουν στην παλιά, άσε που δεν ε, υπάρχει εγγύηση ότι θα επιστρέψουν στην παλιά κατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιστρέψουμε στην κανονική λειτουργία του συστήματος ΣΥΝΚΕΝ και στην εσωτερική αγορά μέχρι τα τέλη του 2016. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν προσβλέπω στις δικές σας απόψεις επί του θέματος και σε προτάσεις για να δούμε πώς μαζί μπορούμε να διασφαλίσουμε τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Επίτροπε. Τώρα, το λόγο θα πάρουν οι εκπροσώποι των πολιτικών ομάδων καταρχήν και πρώτος εκ μέρους του ΕΛΚ, ο κύριος Στάνισλαβ Πόλτσακ. Δύο λεπτά, παρακαλώ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Κύριε Πρόεδρε, λέει ο Πόλτσακ. Κυρίε και κύριοι, αρχίζοντας να σας πω ότι το μεταναστευτικό είναι πρόβλημα κοινό. Είναι πρόβλημα για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και είναι λάθος να ε, θεωρούν ορισμένοι ότι την έχουν γλιτώσει από αυτήν την κρίση. Αυτό είναι λάθος τεράστιο. Και οι συνέπειες του προβλήματος μα αφορούν όλους. Ε, πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα αριθμητικά στοιχεία μα παρέθεσε η Επίτροπο, γι' αυτά προέρχονται από διάφορε ανεξάρτητε μελέτε. Υπάρχουν πάντω κάποιε πολιτικέ ομάδε που τώρα απουσιάζουν από το ημικύκλιο. Είναι ακριβώ εκείνοι οι άνθρωποι που θέλουν το κλείσιμο των συνόρων. Μα εκείνοι θα έπρεπε να ακούσουν τα αριθμητικά αυτά στοιχεία και γενικότερα όλα όσα μα είπε η Επίτροπος, όλα τα οποία ακριβώς αναφέρονται από αυτές τις ανεξάρτητες μελέτες όλα τα σχετικά με το κλείσιμο των σύνορων της ζώνης Σέγγεν. Γιατί ακριβώς ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ελεύθερη διακίνηση και επομένως θα ήταν ε, πάρα πολύ λάθος το να άρουμε αυτή την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, κεφαλαίων, εμπορευμάτων κλπ. Επομένως, η ζώνη Σέγγεν αποτελεί ένα μείζον πλεονέκτημα είναι το κλειδί στην ευημερία και την ανάπτυξη. Ακριβώς λόγω του μεταναστευτικού έχουμε μια απειλή που έχει ε, διαμορφωθεί κατά της ζώνης Σέγγεν. Ακούσαμε ακριβώς πως οι συνδρομικές μεταφορές και οι δικές μεταφορές έχουν ε, χτυπηθεί από την κατάσταση Άρα θα πρέπει να είναι θέμα προτεραιότητα για εμά το να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα και θα πρέπει να είναι σκοπό μα το με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να άρουμε τι ανεπάρκειε που έχουν σχέση με τα σύνορά μα. Και θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί η ζώνη σαν και θα είναι κολοσιαία η ζημία εάν το πρόβλημα δεν επιληθεί. Ακριβώ όπω το είπε κύριε Επίτροπο. Και σα ευχαριστώ, ο Πρόεδρο. Εμεί σα ευχαριστούμε και τώρα για του σοσιαλιστέ, ο κύριο Ισμαήλ Ερτούγκ. Δυόμιση λεπτά. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ξεκινώντας θέλω να διευκρινίσω για άλλη μια φορά ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με μια καθαρή μεταναστευτική κρίση αλλά με μια πολιτική κρίση της Ευρώπης όπως διαπιστώνουμε τους τελευταίους μήνες. Και η κατάσταση είναι η εξής κυρίες και κύριοι, ότι 28 κράτη-μέλη αποτυγχάνουν κατά το τρόπο να δώσουν απάντηση σε μια ανθρωπιστική κρίση η οποία εάν είχε τύχει συντονισμό σε παιδό ευρωπαϊκό με έναν τρόπο λογικό θα είχε βρει λύση πολύ εύκολα. Όσο συντονιστή σοσιαλιστική ομάδα για θέματα των μεταφορών θα περάσω στα θέματα που αφορούν καθαρά τις μεταφορές. Αντί λοιπόν να δοθεί μια συγκεκριμένη λύση, μια ενιαία λύση, άρχισαν ορισμένα κράτη-μέλη να προσπαθούν να πετάξουν το πρόβλημα έξω από την αυλή του. Και έτσι έχουμε να κάνουμε με ένα από τα κύρια προβλήματα που αφορούν το χώρο του Σέγγεν, που κινδυνεύει, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δοθούν λύσεις, του αντίον μάλιστα ε, παρεμποδίζεται η δυνατότητα να μετακινηθούν και να κυκλοφορήσουν ελεύθερα ή 500 εκατομμύρια κάτοικοι με 25 δισεκατομμύρια ταξίδια ανά έτος. Η επαναφορά των ελέγχων στα σύνορα που ανέφερε και ο συνάδελφος επιδεινώνουν και επιμικίνουν τους χρόνους ταξιδιών και άρα και το κόστος. Πληρώνουμε περισσότερα και περιμένουμε για περισσότερη ώρα μέχρι να φτάσουμε στον προορισμό μας. Και για να σας δώσω ένα παράδειγμα κυρία Επίτροπε για τις αρνητικές συνέπειες της ε, επαναφοράς των εθνικών ε, ελέγχων στα σύνορα. Θα σας πω ότι από την επιμελητία υπολογίζεται ότι κάθε ε, ώρα 50 ευρώ για κάθε φορτηγό κοστίσει η μία ώρα αναμονής στα σύνορα σύνορα. Στη γερμανο-αυστριακή μεθόριο, παραδείγματι, έχουμε 8 εκατομμύρια διελεύσεις, 400 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον κόστος δηλαδή. Τέτοιου είδους ε, σκηνικά και σενάρια σημαίνουν δημιουργούν συνέχεια προβλήματα και μπορούν να οδηγήσουν σε 470 δισεκατομμύρια ευρώ απώλεια από το ΑΕΠ μέχρι, μέσα στα επόμενα χρόνια. Παρακαλώ λοιπόν να ε, αναγνωρίσει και η Επιτροπή και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια γιατί μια Ευρώπη χωρίς σύνορα είναι η μόνη Ευρώπη που μπορεί να υπάρχει. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Ερτού. Από την ομάδα ECR τώρα. Κύριος Λοτόφσκι. Έχετε το λόγο, τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, κυρίες και κύριοι. Οι μεταφορές είναι ένα βασικό στοιχείο της οικονομίας μας και η στρέβλωση στις μεταφορές οδηγεί σε οικονομικές απώλειες τους επιχειρηματίες. Συνεπώς, θα οδηγηθούμε και σε απολύσεις στη συνέχεια. Μετά από την μεταναστευτική κρίση λοιπόν, τώρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση χωρίς προηγούμενο για τις μεταφορές. Τα προβλήματα θα είναι πολλά. Εγώ έχω πάρει πάρα πολλά emails από οδηγού από τη δικιά μου προεκλογική περιφέρεια, όπου μου περιγράφουν την κατάσταση που επικρατεί γύρω από το καλέ. Μου αναφέρουν ε, εγκλήματα, ε, τι γίνεται στους δρόμους, πόσο δύσκολο είναι κάτω από αυτές τις συνθήκες να κυκλοφορήσουν τα φορτηγά και φαίνεται ότι η κατάσταση επιδεινώνεται συνεχώς. Έχουμε πολλούς Πολωνούς οδηγούς φορτηγών που αποτελούν ε, την ε, βραχοκοκαλιά του οικονομικού μας συστήματος. Θα ήθελα λοιπόν να μιλήσουμε περισσότερο για την καθημερινότητα των επιχειρηματιών στις μεταφορές και των οδηγών. Έχω δει να πετιούνται πέτρες κατά των φορτηγών και των οδηγών που περνούν στους δρόμους. Ποιος θα αναλάβει το κόστος από τις ζημιές, από τις επισκευές ή από τον έλεγχο που θα πρέπει να γίνεται. Ποιος κινδυνεύει τη ζωή του τελικά. Τραυματίζονται. Ποιος. Οι οδηγοί βέβαια και πλήττονται φυσικά και οι επιχειρηματίες, οι εργοδότες τους και χάνονται πολλά χρήματα καθημερινά. Αυτά είναι κάποια μόνο παραδείγματα του πώς επηρεάζει η μεταναστευτική κρίση των τομέα των μεταφορών. Έπειτα κλείνουν κάποιες δρομικές συνδέσεις μεταξύ χωρών μελών. Τι γίνεται στη Μεσόγειο, άλλο ένα πρόβλημα με πολλές επιπτώσεις, ότι γίνονται με νομερός έλεγχοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα που αντιμετωπίζει ο τομέας των μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι θα συνεχίσουμε και στο μέλλον. Θα κάνουμε κάτι ή θα περιμένουμε να αρχίσουν να χάνουν τη ζωή τους οι φορτηγοί επειδή δεν θα μπορέσουν να μηνθούν, δεν θα καταφέρουν να προστατευτούν από τέτοιου είδου επιθέσεις από τους, μεταναστα... από τους μετανάστες ή επειδή θα είναι εξαντλημένοι στην κούραση. Καλό λοιπόν όλους να βοηθήσουν να χρηματοδοτηθούν επενδύσεις που θα βελτιώσουν την ασφάλεια και την προστασία των οδηγών και όλων όσων αποσχολούνται στις μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε επενδύσει πολλά μέχρι τώρα στις υποδομές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, θα πρέπει να τις προστατεύσουμε αυτές τις υποδομές, να δείξουμε στους πολίτες ποιες είναι οι συνθήκες εργασίες και πώς αυτές επηρεάζονται από τη μετανάστευση. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε ιδιαίτερα τις χώρες εκείνες που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Αν τα εξωτερικά μας σύνορα δεν προστατεύονται επαρκώς, τίποτα δεν θα βοηθήσει. Και ο χώρος Σέγγεν θα διαλυθεί. Το οικονομικό κόστος θα είναι κολοσιαίο και όχι μόνο για τη δικιά μου τη χώρα. Συνεπώς θέλω να κάνω έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητήσω να φροντίσει να επιβληθεί ο νόμος, κάτι το οποίο σήμερα δεν γίνεται. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα εκ μέρους άλλων πολιτικών ομάδων. Ο κύριος Φαν Μίλτεμπορκ έχει τώρα το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η προσφυγική κρίση είναι πάνω απ' όλα ανθρωπιστική κρίση κοστίζει ανθρώπινες ζωές. Και δεν έχουμε όλα τα νούμερα. Και για τις μεταφορές βέβαια υπάρχουν επιπτώσεις. Ως αντίδραση στις μεταναστευτικές κρίσεις, μονομερώς οι χώρες μέλη, κάποιους τουλάχιστον, έχουν κλείσει τα σύνορά τους. Και έτσι εμποδίζουν τη διακίνηση ανθρώπων και εμπορευμάτων. Με μεγάλες επιπτώσεις. Όπως το είπε και η Επίτροπος, επιβεβαιώνει την ε, οικονομική ζημιά με τους υπολογισμούς που έχει κάνει. 5 μέχρι 18 εκατομμύρια το χρόνο μας κοστίζει αυτή η ιστορία και η συστηματική έλεγχη στα σύνορα θα κοστίσουν δισεκατομμύρια. 1,7 έως 7,5 δις το χρόνο επιπλέον κόστος. Αυτή είναι η εκτίμηση. Είναι σαφές λοιπόν ότι πρέπει η αντιμετώπιση να είναι ευρωπαϊκή για να λυθεί το μεταναστευτικό. Με μια πραγματική ευρωπαϊκή συνορφιακή και ακτοφυλακή, με μια πραγματική διαδικασία σύλλου που να εφαρμόσουν όλες οι χώρες μέλη, με την ε, δυνατότητα να υπάρχει νόμιμη μετανάστευση, αλλά και να μην υπάρχουν έλεγχοι στο εσωτερικό του χώρου Σέγγεν. Πρέπει να διαχειριστούμε καλύτερα τη μεταναστευτική κρίση και ανθρωπιστικά, αλλά βοηθώντας και τον τομέα των μεταφορών. Κάνω έκκληση λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να εξακολουθήσει να ερευνά τις επιπτώσεις του μεταναστευτικού στον τομέα των μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζητώ επίσης να μας δώσει νούμερα για τη ζημιά όσον αφορά τα λιμάνια, τους δρόμους, αεροπορικές μεταφορές, πιο συγκεκριμένα και όλα αυτά να έρθει και να τα συζητήσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για να είναι σαφές ότι η Ευρώπη πληρώνει ένα τίμημα επειδή δεν έχει μπορέσει να αντιμετωπίσει την μεταναστευτική κρίση και την έχει αφήσει στις χώρες μέλη. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Εκ μέρους ε, τώρα της ΓΚΟΕ, το λόγο έχει η Τάνια Γκονζάλες Παρακαλώ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας πω για τη ζήτησή μας ότι υπάρχουν πάρα πολλά σημεία τα οποία με βρίσκουν σύμφωνοι αλλά και άλλα τα οποία με ανησυχούν γιατί νομίζω ότι είναι απαραίτητο να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ε, το μεταναστευτικό αλλά σε πολυεπίπεδα και πολλέ απόψεις για να μπορέσουμε να βρούμε αποτελεσματικές και βιώσιμες ε, λύσεις μέσω και μακροπρόθεσμες πρώτα απ' να τονώσουμε το τι γίνεται ε, με τα σκάφη εκείνα τα οποία διασώζουν τα σκάφη τα οποία έχουν παρασυρθεί από τα κύματα στις θάλασσές μας. Επίσης ε, έχουμε ε, τον ΟΗΕ που θεωρεί ότι η Μεσόγειος είναι πιο θανάσιμη οδός για τις μεταναστευτικές ροές και θα πρέπει να δούμε πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η, δορυφορική τεχνολογία. Οπότε έτσι είναι δυνατόν να υπάρχει εντοπισμός, να υπάρχει βοήθεια και αυτό βέβαια θέλει και κάποιο προετοιμασία. Πρέπει να δούμε επίσης τι θα γίνει με κάποιες κυρώσεις που υπάρχουν ε, και από επιχειρήσει αλλά και από το κράτος όταν τα σκάφη αυτά πιάνουν λιμάνι. Θα πρέπει μέσα στα κράτη-μέλη να κάνουν κάποιες επιχειρήσεις διάσωσης ανθρωπιστικές. Θα πρέπει επίσης τα εμπορικά σκάφη να έχουν τα ε, πληρώματα, πρωτόκολλα κατάρτισης και εκπαίδευσης. Πάντως, εκτός από όλα αυτά υπάρχουν κάποια σημεία που με ανησυχούν. Γιατί στο επίκεντρο της προβληματικής έχουμε αποκλειστικά θέματα σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα και με την εύρεθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Ε, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι αυτά τα θέματα είναι πολύ σημαντικά για μας. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το πιο ενισχυτικό. Το ότι έχουμε ολοένα και περισσότερες μαφίες που διακινούν τους ε, μετανάστες ε, και τους ζητάνε για να τους μεταφέρουν χίλια ευρώ για παράδειγμα και τους βάζουν σε ένα φορτηγό ενώ έχουν αλληλεγγύες λύσεις που είναι πιο φτηνές αλλά ο κοσμάκης αυτός δεν έχει ιδέα, κανείς δεν τους ενημερώνει. Άρα θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτούς που εκμεταλλεύονται τον απελπισμό, την, την, την απελπισία τους και να μην τους γυρίζουμε την πλάτη όταν έχουμε τόσα θύματα. Πολλοί πεθαίνουν ε, από ασφυξία. Ε, α, τις προάλλες αυτό έγινε. Μέσα σε ένα φορτηγό ε, ψυγείο στην Αυστρία βρέθηκαν νεκροί μετανάστες οπότε ή πρόκειται για θέμα το οποίο με κάνει να νιώσω ντροπή. Επίσης θα πρέπει να, είπαμε, να, να, να λειτουργεί εύρεθμα η ζώνη Σέγγεν. Μα αφού η, η ροή, η, η ανεμπόδιστη και η ελεύθερη ε, κυκλοφορία μας, ε, μας ενδιαφέρει γιατί τότε να μην κάνουμε κάτι για το Ενωμένο Βασίλειο το οποίο βάζει τόσες ε, τροχοπέδες στην ελεύθερη διακίνηση. Είναι δικές μας ευθύνες όλα αυτά. Καθόμαστε και είμαστε θεατές και δεν κάνουμε τίποτα. Θα πρέπει να, η Υπουργή να είναι δημοκρατική και να βάζει στο επίκεντρο τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος προς την κυρία Γκονθάλεφ Πένιας. Και... Τώρα εκ μέρους των Πρασίνων η κυρία Καρυμαντελή. Δύο λεπτά παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλούμεθα να συζητήσουμε τι συνέπειε μεταναστευτική, τη κρίση των προσφύγων στον τομέα των μεταφορών τη Ευρώπη. Ξεκινώντα, θέλω να σα πω ότι διατύπωση αυτή με ενοχλεί βαθύτατα. Από τον Ιούνιο του 2015 έχουμε, πάνω, έχουμε 9 νεκρούς ε, στο τούνελ ε, του, της μάχης. 70 τον Ιούνιο του 2015 σε ψυγείο φορτηγό στην Αυστρία. Δεν έφταγαν εκεί οι μεταφορές, όπως και δεν έφταγαν στο τούνελ της μάχης. Στη Μεσόγειο, 4.000 νεκροί το χρόνο από το 2014. Πάλι δεν είναι ε, υπέτειες οι θαλάσσιες μεταφορές. Γι' αυτό λοιπόν μερικές φορές βρίσκουμε στην ομάδα ε ΕΝΕΛ την ρητορική αυτή που θέλει να ρίξει όλα τα φταξίματα στους πρόσφυγες. Η Κυρνία Αρναουτού την προηγούμενη εβδομάδα από το Front National υπέβαλε πρώτη στην Επιτροπή των Μεταφορών μια, μια πρόταση λοιπόν για τις ακτοφυλακές, συνοριοφυλακές όπου μας λέει πως η κρίση των προσφύγων οδηγεί στο ε, δυσάρεστο, στη δυσάρεστη συνέπεια να αναγκάζονται και παραθέτω τα λόγια της ε, κάποια σκάφη του εμπορικού ναυτικού να αλλάζουν ρότα για να συμμετάσχουν σε ε, εργασίες διάσωσης. Μα δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να χτυπήσουμε τους λαθροδιακινητές, να βρούμε λύσεις για την σύγκρουση στη Συρία, αλλά πάνω απ' όλα να καταγγείλουμε την ανικανότητα των κρατών και των κυβερνήσεων να δώσουν απαντήσεις σε όλα αυτά τα προβλήματα και σε όλους εδώ τους συναδέλφους θέλω να πω ότι δεν μπορούμε να δώσουμε απάντηση αξιοπρεπή στην κρίση εάν δεν έχουμε κάνει ό,τι περνάει από το χέρι μας για να δώσουμε απαντήσεις. Στη δική μου την περιοχή, στην Grand ο δήμαρχος Ντανιέλ Καρέμ έχει εγκαταστήσει καταβλισμό που υποδέχεται σε όρους αξιοπρέπειας τους πρόσφυγες, ενώ αλλού στη Βουλγαρία, παραδείγματι, ε, Του έρνουν σιδηροδέσμιου ε, στην Αυστρία επί παραδείγματι προσπαθούν να σκαρφαλώσουν τύχη είναι όνειρο αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ευθύνη κοινή όλων μας είναι και οι λέξεις που θα διαλέξουμε και οι πολιτικές μας επιλογές και οι πράξεις μας Α σταματήσουμε λοιπόν να χρεώνουμε όλα τα φταξίματα στου πρόσφυγε. Ευχαριστώ πολύ κύριε, ε, κυρία Τελή Δεν βλέπω τον κύριο Μάιερ εδώ. Μάλλον απουσιάζει. Μεγέχ. Η κυρία Μορβάη όμω είναι εδώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εξήμιση χρόνια τώρα βρίσκομαι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και νομίζω ότι έχω αρχίσει να καταλαβαίνω την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μην με παρεξηγείτε. Δεν εννοώ ότι διανοητικά έχω αλλάξει. Αυτό που λέω είναι ότι έμαθα τα κόλπα σας, τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεστε, τον τρόπο με τον οποίο προσπαθείτε να πουλήσετε τις περίεργες ιδέες σας στον κόσμο. μέσω των δικών σας ανατρεπτικών μέσων. Κοιτάξτε, είναι εδώ η Επίτροπος για να μας πει φοβερά πράγματα για το πόσο πολύ κοστίζει η επενισαγωγή των ελέγχων στα εσωτερικά σύνολα, σύνορα εξαιτίας του μεταναστευτικού και ότι γι' αυτό κοστίζει πολλά χρήματα στον Ευρωπαίο φορολογούμενο. Ε, εντάξει, μα τι πρέπει να κάνουμε, να σταματήσουμε τη μαζική μετανάστευση. Αλλά δεν είναι αυτό που προτείνεται. Οπότε περιμένουμε μέχρι την επόμενη φορά. Θα αφήσουμε με νόμιμη μετανάστευση να μπουν όλοι μέσα. Αλλά ακόμα και αυτό θα ήταν εντάξει, συνάδελφοι, εφόσον οι χώρες οι οποίες θέλουν να υποδεχτούν μετανάστευση, να τους υποδεχτούν και οι άλλες που δεν θέλουν να μην τους υποδεχτούν. Αλλά δεν κάνετε αυτό. Αυτό που κάνετε είναι ότι προσπαθείτε να υποχρεώσετε και την ε, Ουγγαρία και να την στριμώξετε. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, δέχεστε μία μπλε κάρτα από τον κύριο Πολτσακ. Ναι. Ευχαριστώ. Θέλω. Ναι, δεν είμαι εγώ σαν τον Άλμπρεχτ και τους κακούς των φιλελευθέρων. Εγώ δέχομαι ερωτήσεις και ακόμα και από τους πολιτικούς μου αντιπάλους. Μάλιστα. Κύριε Πόλτσακ, έχετε το λόγο για 30 δεύτερα. Επιθυμίζω ε, 30. Ευχαριστώ πολύ κυρία συνάδελφε που δεχθήκατε την ε, μπλε κάρτα. Ε, δεν μπορώ να διαφωνήσω περισσότερο με την κυρία Μορβάη. Και έτσι δεν μπορούσα να κρατηθώ και να υποβάλω την εξερώτηση. Εσείς τη δήλωση ότι το να κλείσουν τα σύνορα του Σέγγεν δεν πρόκειται να φέρει επιπτώσεις στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πού τη στηρίζετε. Γιατί δεν ρωτάτε την Επιτροπή, ε, γιατί αφού εσείς ρωτάτε την Επιτροπή από πού αντλεί τα στοιχεία της, δεν μας λέτε τα δικά σας τα στοιχεία, κυρία Μορβάη. Είμαι ιδιαίτερο ευγνώμων για την ερώτηση, γιατί φαίνεται ότι προφανώς δεν ήταν κατάλληλη η μετάφραση και θα σας τα πω στα αγγλικά για να με καταλάβετε. Προφανώς συμφωνώ ότι υπάρχει τεράστιο κόστος από το κλείσιμο των εσωτερικών συνόρων και για την για τους ε, συμπολίτε μου, τους συμπατριώτες μου, τους Ούγκρους, αλλά η απάντηση θα πρέπει να είναι να σταματήσουν οι μαζικές μεταναστευτικές ροές. Ωστόσο αυτό δεν πρόκειται να το πράξετε. Η σημερινή συνεδρίαση ήταν μια προετοιμασία για μια επόμενη και μεθεπόμενη στην οποία θα ανακοινώσετε πως θα πρέπει να καταστεί νόμιμη κάθε μορφή μετανάστευσης που εμείς οι Ούγγροι δεν θέλουμε και δεν μπορείτε να μας την επιβάλλετε. Αυτό είχα να πω και ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, αγαπητοί συνάδελφοι. 30 δεύτερα υπενθυμίζω για την ερώτηση και 30 δεύτερα για την απάντηση επίσης. Άντορ Ντέλη, δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το θέμα δεν είναι μόνο η κρίση και τα προβλήματα ανταγωνιστικότητας που φοβούνται και έχουν αντιμετωπίσει τώρα εταιρείε μεταφορών, αλλά το μεταναστευτικό μα οδηγήσει σε όλο ένα περισσότερου μεθοριακού ελέγχου και έτσι έχουμε όλο ένα και λιγότερα εμπορεύματα να καταλήγουν εκεί που πρέπει. Και βέβαια έχουμε και αύξηση του κόστους και σε ιδιαίτερα μεγάλες χρονικές περιόδους. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα για τα ευαίσθητα προϊόντα. Ε, πάρα πολύ επιβάτες ε, χάνουν το χρόνο τους, αλλά επιβαρύνεται και το περιβάλλον επομένως θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τις τέσσερις βασικές ελευθερίες και την ενιαία αγορά να μπορέσει να λειτουργήσει ε, το σύστημα Σέγγεν, ζώνη Σέγγεν σύμφωνα με τους ε, κανόνες πρέπει να ενεργοποιηθούν πλήρως. Επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το τι θα γίνει ε, με το επάγγελμα των οδηγών των φορτηγών. Είναι η δουλειά τους και όλο ένα και περισσότερα προβλήματα αντιμετωπίζουν, άρα για κινδύνους Άρα θα πρέπει να τους ασφαλίσουμε ασφαλείς συνθήκες εργασίας. Είναι πολύ σημαντικό για εκείνους. Και έχουμε την οδηγία 89 και 391 θα πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως. Αλλά επίσης θα πρέπει να φροντίσουμε το δίκτυο, θα πρέπει γενικά να προστατεύσουμε την υγεία των οδηγών των φορτηγών. Αλλά να μην ξεχνάμε για τον τουρισμό, διότι οι τρομοκρατικές επιθέσεις ε, και οι τρομοκρατικές ε, απειλές έχουν πλήξει τον τουρισμό. Μην ξεχνάτε ότι ο τουρισμό το 10% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ είναι πολύ σημαντικό κλάδο. Επομένω, οι εκεί οι ζημίες ε, έχουν χτυπήσει πολύ σοβαρά την οικονομία μα. άρα θα πρέπει να δούμε το πώ θα μπορέσουμε να αντισταθμίσουμε τι ε, τις αυτέ ε, ζημίες αυτές από τον τουρισμό, αλλά και από τις μεταφορές. Θα πρέπει κάτι να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ε, ξαλαφρώσει το βάρος από τη ζημία. Ευχαριστούμε λέει ο Τώρα η κυρία Αγιάλα Σάντερ. Δύο λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Διαπιστώνουμε και πάλι το τίμο πρέπει να πληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτία ενό ιστορικού σφάλματο έλλειψης συντονισμού των πολιτικών μας. Και επειδή υπερισχύουν οι εθνικοί εγωισμοί, όλα αυτά συνδυασμένα είναι σε βάρο των πολιτών μα δεν υπάρχει πολιτική, είναι λανθασμένη η <clears throat> διακυβερνητική και αυτή είναι που έχει οδηγήσει στους εγωισμούς σε βάρος των μεταναστών και των προσφύγων. Με ε, ένα κόστος πολύ μεγάλο. Το Σέγγεν είναι μέρος της Ευρώπης αυτής, πιο ενωμένης όπως τη θέλουμε. Έτσι λοιπόν κύριε Επίτροπε, στηρίζουμε την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διατηρήσει το Σέγγεν και θα αγωνιστούμε ώστε όσο γίνεται πιο γρήγορα να είναι και πάλι ανοιχτά όλα τα σύνορα στην Ευρώπη. Συγχρόνως θέλουμε να βρούμε καλύτερους τρόπους ανθρωπιστικής διαχείρισης των μεταναστών και όσου ζητούν άσυλο σε εμά που προσπαθούν να ξεφύγουν από τα βασανιστήρια και τον πόλεμο στις χώρες τους. Οι μεταφορές πλήττονται θα μπορούσαμε να είχαμε ασφαλείς ανθρωπιστικούς διαδρόμους. Αυτό το έχουμε ζητήσει από την αρχή. Τότε οι μεταφορές θα μπορούσαν να ήταν η λύση για να αποφεύγουμε θανάτους. Μια ανθρωπιστική εναέρια γέφυρα από την Ελλάδα επίσης προς τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες θα μπορούσαν να πάρουν πρόσφυγες και μετανάστες. Και αυτό θα είχε βελτιώσει πάρα πολύ τη σημερινή κατάσταση. Ενώ ανταυτού έχουμε κατακαιρματισμένες λύσεις, λανθασμένες. Πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Όσο γίνεται πιο γρήγορα να ανοίξουμε τα σύνορα, να έχουμε συντονισμένα μέτρα για να διευκολύνουμε την μεταφορά και να ενισχύσουμε έτσι τους εργαζόμενους στον τομέα των μεταφορών. Οι εθνικές κυβερνήσεις βάζουν και υιοθετούν δικά τους μέτρα χωρίς να είναι σε συντονισμό με την υπόλοιπη Ευρώπη πρέπει να μην συνεχίσουμε να κάνουμε τα ίδια σφάλματα, να το πούμε αυτό στο Συμβούλιο. Ελπίζω η επίτροπο να μπορέσει να βοηθήσει. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε μια εσωτερική αγορά και τα ανθρώπινα δικαιώματα έτσι όπω τα θέλουμε με κλειστά τα σύνορά μα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ κύριε Γαλασέντερ. Τώρα. Ο κύριος Άγγελ Νταμπάσκι έχει το λόγο. 1,5 λεπτό κυβέρνηση του Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Η κυρία Τάισεν, κοιτάξτε, συζητάμε σήμερα ξανά για τη μετανάστευση. Και έχω την αίσθηση ότι μιλάμε διαφορετική γλώσσα παρόλο που έχουμε διερμηνία στη διάθεσή μας. Γιατί μερικοί συνάδελφοι δεν κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Και μετά τους εκπλήσει όταν διαπιστώνουμε ότι έχουμε τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι, στις Βρυξέλλες. Αυτή η μεταναστευτική κρίση επηρεάζει πάρα πολύ τον τομέα των μεταφορών. Οι διεθνείς μεταφορές ξέρουν ότι αν συνεχιστεί η μεταναστευτική κρίση, οι έλεγχοι θα γίνουν ακόμα πιο αυστηροί και το αποτέλεσμα θα είναι να χάσουμε εκατομμύρια και εκατομμύρια στον τομέα των μεταφορών. 5 με 18 δισεκατομμύρια εκτιμάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα είναι η απώλεια. Ε, βέβαια, θα αποθαρρυνθεί ο κόσμο να ταξιδεύει στην Ευρώπη. Για να διατηρήσουμε λοιπόν το Σέγγεν και τη λειτουργία τη εσωτερική αγορά, θα έπρεπε να ενισχύσουμε του ελέγχου στα σύνορά μα. Στη Βουλγαρία, για παράδειγμα. Μην είμαστε υποκριτέ. Δεν είναι δυνατόν μερικοί να είναι κομμάτι του Σέγγεν και άλλοι να μην είναι. Εμεί δεν θέλουμε να είμαστε στο Σέγγεν, γιατί δεν πρόκειται να έχουμε πλέον εκτίματα από το να είμαστε στο Σέγγεν. Από την άλλη μεριά όμω η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει συμφωνίε με την Τουρκία και ζητάμε από την Τουρκία να προστατεύσει τα δικό μα ε, σύνορα. Ανοίγουμε την ε, πόρτα επίση στα τουρκικά να γίνουν επίσημη γλώσσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι μέγα σφάλμα. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Νταμπάσκη. Η κυρία Ινές Γιάλα Σάντερ, που μίλησε πριν από εσά, έχει μία μπλε κάρτα. Θέλει κάτι να σας ρωτήσει πάνω στις διαδικασίες της μπλε κάρτας. Συμφωνείτε από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, παρακαλώ, κυρία Γιάλα Σάντερ, ακόμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την κατανόησή σας. Θέλω να υπενθυμίσω στον Ευρωβουλευτή ότι οι τρομοκράτες δεν ήταν ούτε μετανάστες, ούτε πρόσφυγες, ήταν Ευρωπαίοι πολίτε Οπότε λάθος κάνετε. Απάντηση. Ε, αυτή δεν είναι ερώτηση που κάνατε, ήταν μια δήλωση. Οπότε παραβιάζετε τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρ' όλα αυτά θα σας δώσω μια απάντηση. Ελάτε στα σύνορα Βουλγαρίας-Τουρκίας και δείτε τα από μόνοι σας ποιος είναι πρόσφυγας και ποιος είναι παράνομος μετανάστης. Λένε 30χρονοι νέοι άντρες ότι είναι το ίδιο με γυναίκες με παιδιά. Ε, δεν είναι, δεν έχετε δίκιο. Ελάτε στα σύνορα αυτά να δείτε την κατάσταση από μόνοι σας. Ευχαριστούμε. Τώρα το λόγο έχει η κυρία Μπιλμπάο Μπαραντικά. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε ποιε είναι οι ανθρωπιστικέ συνέπειε αλλά και οι πολιτικέ για την Ευρώπη από το προσφυγικό. Θα, το ότι θα πρέπει ε, τώρα να έχουμε καινούργιου ελέγχου αυτό πρόκειται να προσθέσει 18 εκατομμύρια ε, όπως λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άρα θα πρέπει να δώσουμε τριπλάσιους πόρους για την Τουρκία στα πλαίσια της συμφωνίας και θα έχουμε επίσης και κάποιες επενδύσεις στα δικτύα ώστε να υπάρχει αποδοτικότητα ε, με όλους αυτούς τους ελέγχους. Αυτό κοστίζει το 1% του ΑΕΠ. Οπότε επί τη βάση αυτών σας ερωτώ τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εμποδίσει λαϊκιστικά μονόπλευρα μέτρα κατά της ευθές διακίνησης προσώπων και εμπορευμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά δεύτερον, τι μέτρα μπορείτε να πάρετε τόσο ώστε να αντισταθμίσετε αυτό το κόστος που θα χτυπήσουν την ανταγωνιστικότητα ε, όλων των οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρόεδρος, ευχαριστούμε εμείς, κυρία. Και τώρα η κυρία Μαρή Κριστίν Βερζιότ, δύο λεπτά. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, μπράβο που προσπαθείτε να μιλήσετε σε όλες μας τις γλώσσες. Ναι, το, το, το, το εμπόριο ε, πολλά από εμπορικά πλοία που υπάρχει και πάνω από 800 έχουν σώσει στην ε, Μεσόγειο τα εμπορικά πλοία και αυτό πρέπει να χαιρετιστεί γιατί κάνα το κάθε οίκον τους παρά όλα τα εμπόδια σύμφωνα με το δίκαιο. Είπαμε ότι όλο και περισσότερα τέτοια πλοία αλλάζουν ε, την πορεία τους, τόσο ώστε να ε, μην ε, μπαίνουν στα δρομολόγια των μεταναστών. αυτών των μεγάλο πρόβλημα. Και έχουμε 30.000 νεκρούς από το 2002 και 3.700. Αυτό είναι ένα κόρο, οπότε ναι, έχει γίνει η πιο θανάσιμη περιοχή για τους μετανάστες, η Μεσόγειος το 2014 ήταν πρώτη η Ιταλία, είχαμε 5 εκατομμύρια τα οποία είχαν διαθέσει και, και άλλα 95. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τους διακινητές, πώς θα είναι δυνατόν να ε, σταθμίσουν το κόστος γιατί στρατεύεται ε, και ο στρατός οπότε θα πρέπει να δούμε το ότι κοστίζει ολένα ένα περισσότερο και ολένα ένα περισσότερου κινδύνου επιφυλάσσει αυτή η διακίνηση των μεταναστών. Είναι τώρα με τα ναρκωτικά και όπλα για αυτές τις συμμορίες είναι η τρίτη πηγή κέρδους. Και όσο πιο πολύ κλείνουν τα σύνορα, τόσο πιο πολύ ανθούν αυτές οι επιχείρησεις. Είχαμε τεράστιο κόστος από το κλείσιμο των σύνορων. Τόσα χρήματα θα μπορούσαν να σώσουν ζωές επί τη βάση του διεθνούς δικαίου τα δικαιώματα να προστατεύσουν μεταναστών και προσφύγων. Άρα θα πρέπει η Ένωση να βοηθήσει αυτήν την ανθρωπιστική κρίση που λάβαμε λοιπόν, στα μάτια μας. Θα πρέπει να έχουμε κοινοτική μεγάλη εμβέλεια επιχείρηση για να σώσουμε ζωές, να ανοίξουμε ανθρωπιστικούς διαδρόμους και να επίσης ανοίξουμε νόμιμες οδούς μετανάστευση στον κόσμο. Αυτά επί τη βάση του δικαίου και του κοινωτικού δικαίου, οπότε να μην χρειαστεί να τα ξανασυζητήσουμε αυτά. Ευχαριστούμε κυρία Βερζιά, λέει ο πρόεδρος. Και τώρα ο κύριος Πόσπισιλ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Τίσεν για τις ε, πληροφορίες αυτές με τις οποίες ε, ταυτίζομαι διότι θεωρώ ότι η κατάργηση του Σέγγεν θα οδηγούσε σε πολλά προβλήματα όχι μόνο εμάς αλλά και άλλες χώρες. Για δε τις μεταφορές θα σήμαινε απώλεια 500 εκατομμύριων ευρώ κατέτος εάν ε, αποκατασταθούν τα ιστορικά σύνορα. Και δυστυχώς είναι πραγματικά τα στοιχεία αυτά. Ιδιαίτερα για εκείνους που ζουν στην παραμεθόρο και εργάζονται από την άλλη πλευρά των συνόρων, ε, θα δυσκολέψει πολύ και η, δουλειά, και η ζωή και ο επαγγελματικός βίος. Στα ταξίδια, στον τουρισμό, στην αναψυχή θα έχουμε συνέπειες οικονομικές αλλά και γενικότερα στην ευημερία των συμπολιτών μας, γιατί θα ήταν πολύ πιο περιορισμένοι στην να ταξιδεύουμε. Έχουμε λοιπόν στοιχεία που δείχνουν ότι το Σέγγεν έχει μεγάλη σημασία. Παρότι φαίνεται ότι πολλοί Ευρωπαίοι σήμερα δεν φαίνεται να το πιστεύουν και δηλώνουν ότι θέλουν να αποκατασταθούν τα ιστορικά σύνορα. Αυτό δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει διαχειριστεί σωστά την προσφυγική κρίση. Κυρία Τέσσιν, πιστεύω, θα πρέπει από πλευρά τη να αντιληφθεί ότι είναι σημαντικό το Σέγγεν και άρα χρειάζεται να ληφθούν μέτρα για να αντιμετωπιστεί η κρίση και νομίζω ότι εάν ε, εισαχθούν ποσοστώσεις προσφύγων η κοινή γνώμη θα αντιδράσει πολύ αρνητικά και θα αμφισβητήσει και πάλι το Σέγγεν. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ασής παρακαλώ. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η μερική άρση λειτουργίας του συστήματος Σέγγεν είχε σημαντικές συνέπειες και είναι ξεκάθαρο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει την προσφυγική κρίση. Και όταν λέω Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εννοώ Επιτροπή. Γιατί η Επιτροπή προσπάθησε με μια σειρά μέτρων να δώσει απαντήσει στην προσφυγική κρίση. Και αυτό δεν μπορούμε να το αγνούμε. Πρόβλημα όμως ε, υπάρχει ως προς τη συμπεριφορά ορισμένων κρατών μελών. Είδαμε πρόσφατα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη να εισάγουν μέτρα που παραβιάζουν ξεκάθαρα το πνεύμα του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Κράτη με, αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων μιλούν ε, με ορολογία που αποκλείει τον ε, έτερο, μερικές φορές ε, χρησιμοποιούν ρητορική ξενοφοβική ακόμη και βλέπουμε να προσπαθούν να αναιρέσουν τους ε, όρους λειτουργίας του Σέγγεν που όμως έχει κρίσιμη σημασία, ζωτική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί μια από τις κύριες αρχές της ε, Ένωσης είναι η ελεύθερη διακίνηση. Πέραν των αρνητικών οικονομικών επιτάσεων θα πρέπει να εξετάσουμε και τις γενικότερες συνέπειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κινδυνεύει η ίδια η ψυχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τέτοιου είδους περιφορές και όπως είπαν οι άλλοι να για να αναφέρω και εγώ οικονομικά στοιχεία βεβαίως θα είναι πολύ σοβαρές οι επιπτώσεις σε οικονομικούς όρους Πρέπει πάντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την παρακαλώ να απευθύνει διαρκώς εκκλήσεις προς τα κράτη-μέλη για να τηρήσουν τους όρους του Σέγγεν. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος, τον κύριο Ασής. Και τώρα... Η κυρία Άγνες Κιονκέριος. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, την προηγούμενη εβδομάδα ήμουνα με ένα φορτηγό Ολλανδικό στην, ε, προς την Αγγλία. Τη νύχτα. Και ήταν εντυπωσιακό. Γιατί περάσαμε από το καλέ, αλλά δεν μπορώ να πω ότι αισθανόμουν ασφαλής παρά το ξεκαθάρισμα που έχει γίνει υποτίθεται εκεί. Και κάπου κοντά στα γαλλικά ε, σύνορα είδαμε τους μετανάστες εκεί και υπήρξαν και κάποια επεισόδια. Το Μάρτιο βρέθηκαν κάποιοι κρυμμένοι στα φορτηγά να περνάνε από το καλέ και συνεχίζονται τέτοια επεισόδια. Η Επιτροπή λέει ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις οικονομικές επιπτώσεις του κλεισίματος των συνόρων. Ναι, αλλά πρέπει να δώσουμε περισσότερη σημασία και στη συνεργασία στην Ευρώπη. Καλύτερη καταγραφή και καλύτερη προστασία των επιχειρηματιών που εργάζονται στον τομέα των μεταφορών. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γιονγκέριους. Και τώρα αρχίζει η διαδικασία Catch the Συν Κέλλη είναι ο πρώτος που έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε διάφορα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι μεταφορές σε σχέση με την μετανάστευση. Δεν είχα αντιληφθεί όμως ότι ήταν τόσο άσχημα τα πράγματα όπως μας είπατε. Άκουσα τα νούμερα, είναι κάπως ασαφή. Όταν λέτε 5 με 18 δισεκατομμύρια, μα είναι πιο πολύ στο 5 ή πιο πολύ στο 18. Η διαφορά είναι τεράστια, θα έπρεπε να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Πάντως έτσι καλώ είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα και έχοντας μιλήσει με διάφορους με διάφορους οδηγούς φορτηγών με τους οποίους μάλιστα θα φάω και το βράδυ ξέρω ότι η κίνδυνη είναι μεγάλη. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση υπέρ των δικών μας ανθρώπων, των Ευρωπαίων που χρησιμοποιούν τις μεταφορές. Η Επιτροπή λοιπόν πρέπει να προσπαθήσει να βρει έναν τρόπο για νόμιμη μετανάστευση. Γιατί αν δεν υπάρχει νόμιμη μετανάστευση δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Γιατί όταν κάτι είναι παράνομο όλα επιτρέπονται. Ελπίζω οι χώρες μέλη να συνεργαστούν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Λέω ο ο κύριος Μάμικιντς έχει τώρα τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, τι συζητάμε εδώ σήμερα. Συζητάμε το εξή. Η μεταναστευτική κρίση έχει επιπτώσει στον τομέα των μεταφορών. Η μεταναστευτική κρίση θα έχει επιπτώσει σε όλους τους τομείς, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Οικοδόμημα. Αν αναλύσουμε τις αιτίες, γιατί δηλαδή η μεταναστευτική κρίση είναι τόσο μεγάλη και γιατί έχει φτάσει στα σπίτια μας, μία είναι η απάντηση έχουν γίνει τεράστια σφάλματα στην εξωτερική μας πολιτική. Και εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση τα πράξαμε τα σφάλματα αυτά, αλλά και κάθε χώρα χωριστά με τις δικές της αποφάσεις τα τελευταία χρόνια. Οι μετανάστες έρχονται από αυτές τις χώρες στις οποίες εμείς οι Ευρωπαίοι, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινεί με τους ε, εαυτούς μας, τους φέραμε. Δεν έρχονται από πουθενά οι μετανάστες έρχονται για να ζητήσουν τη δικιά μας βοήθεια. Και αυτό είναι που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ιβαρ Βιάκοβιτς. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τις ευκαιρίες να μιλήσω και προς άλλους συναδέλφους από τους φιλελευθέρους. Ναι, ευχαριστώ. Είχατε πει από την αρχή. Τώρα εντάξει. Λοιπόν, το Σέγγερ είναι από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι απλώς διευκόλυνση στο να περνάμε τα σύνορα λιγότερες ουρές και απουσία ουράς. Πολλά περισσότερα είναι. Είναι ένα σύμβολο το Σέγγεν και γι' αυτό πρέπει να το διαφυλάξουμε. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το προστατέψουμε. Η μεταναστευτική κρίση είναι μια τεράστια πρόκληση. Δεν θα είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί, το ξέρουμε πολύ καλά. αλλά πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε και αυτό το απευθύνω σαν έκκληση προς την Επίτροπο και τα κράτη-μέλη για να διασωθεί το Σέγγεν. Ευχαριστώ πολύ. Από την ίδια... Από την ίδια ομάδα, κύριο κύριος Πρόεδρε, ευχαριστώ. Μιλάμε για σύνορα, Σέγγεν, μεταναστευτική κρίση. η Μεσόγειος έχει μετατραπεί σε ένα νεκροταφείο, καθώς οι άνθρωποι προσπαθούν να βρουν παράνομους τρόπους, πέφτουν στα χέρια των λαθροδιακινητών και της μαφίας για να περάσουν στην Ευρώπη. Δεν πρέπει να λησμονήσουμε ότι τα μεσογειακά σύνορα, η Μεσόγειος, είναι εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν μπορεί να κλείσει με, με τύχη, όπως νομίζουν κάποιοι ότι σε άλλα μέρη της Ευρώπης μπορούν να ορθώσουν. Τα σκάφη βρισκόνται στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωση Από την αρχή του χρόνου το 1 τρίτο των μεταναστών ε, που διασώθηκαν στη θάλασσα διασώθηκαν από εμπορικά σκάφη. Δεν θα έπρεπε λοιπόν κύριε Επίτροπε να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ε, αντιμετώπιση κατά τρόπο αποτελεσματικό του θέματος ασφάλειας στη θάλασσα. Δεν θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ε, θαλασσιών μεταφορών να αναβαθμιστεί. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα παρακαλώ την Επίτροπο, κυρία Τάισεν, να λάβει το λόγο. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πολύ για την ανταλλαγή αυτή απόψεων. Σας ευχαριστώ πολύ για τις απόψεις και τις σκέψεις σας. Πράγματι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολείται πολύ και είναι προτερότητά της η αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης. Να κάνουμε δηλαδή ό,τι περνάει από τα χέρια μας για να αποφύγουμε και την τρομοκρατία. Αλλά εδώ συζητάμε για τις επιπτώσεις της μεταναστευτικής κρίσης στον τομέα των μεταφορών. Ας περιοριστούμε λοιπόν σε αυτή τη συζήτηση. Ας επικεντρωθούμε σε αυτό. Η έλεγχοι στα σύνορα είναι σαφές ότι πρέπει να είναι προσωρινή και το αργότερο, το εντελώς αργότερο θα πρέπει να έχουν σταματήσει στα τέλη της χρονιάς, μετά δηλαδή από 8 μήνες. Είπα στην αρχή το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που σας παρουσίασα 4 Μαρτίου ότι υπάρχει προκειμένου να επανέλθουμε στην κανονική λειτουργία του χώρου Σέγγεν. Υπάρχει ανακοίνωση της Επιτροπής. Αυτό θέλουμε και αυτό σας έχουμε παρουσιάσει ξέροντας ότι ο χώρος Σέγγεν είναι μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επανέλθουμε στην κανονική λειτουργία του Σέγγεν. Αυτό είναι που θέλουμε Αυτά λέει και η ανακοίνωση και πράγματι το κόστος από την έλλειψη του Σέγγεν είναι τεράστιο από πολλές απόψεις γιατί και την ελευθερία μας πλήττει αλλά και οικονομικό είναι το κόστος. Στόχος μας λοιπόν είναι όσο γίνεται πιο γρήγορα να επανέλθουμε στην πραγματικότητα και στην προηγούμενη κατάσταση. Όσο γίνεται πιο γρήγορα να λειτουργήσει κανονικά το Σέγγεν για να επωφελούμεθα από τα πλεονεκτήματά του. Πρέπει να φροντίσουν οι χώρες μέλη λοιπόν να γίνει αυτό πραγματικότητα. Τώρα λέτε να παρακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την κατάσταση, το κάνει και στα εσωτερικά σύνορα και στα εξωτερικά σύνορα και όντως εκτιμήσεις έχουμε για το κόστος προς το παρόν, γι' αυτό σας έδωσα τα ποσά αυτά. Μπορεί να ακούγονται μεγάλα τα ποσά, είναι σιγά σιγά αναλύοντας περισσότερο ε, την κατάσταση και τα στοιχεία που έχουμε θα μπορούμε να είμαστε περισσότερο πλήρεις για το κόστος της κατάστασης αυτής. Πάντως το κόστος θα είναι μεγάλο. Γι' αυτό και θέλουμε να επανέλθουμε στην κανονική λειτουργία του Σέγγεν. Και το κόστος θα είναι μεγάλο για τις μεταφορές, για τις χώρες μέλη. Όλους μας πλήττει αυτή η κατάσταση, όχι μόνο τις μεταφορές. Αν γυρνάμε την πλάτη στο Σέγγεν και στα πλονεκτήματά του, τότε το κόστος θα είναι τεράστιος για ολόκληρη την οικονομία μας, για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και για την ε, λειτουργία των συνόρων. Συνεπώς, έχω εμπιστοσύνη ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε όπως χρειάζεται ώστε να αντιμετωπίσουμε την κρίση αυτή και να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε πλήρως την εσωτερική μας αγορά για τις μεταφορές και να έχουμε την ελεύθερη διακίνηση ατόμων και εμπορευμάτων, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την οικονομία μας ολόκληρη. Σας διαβεβαιώ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όλοι οι επίτροποι, κυρίως ο Επίτροπος Αρμόδιος για τις Μεταφορές, όλοι είμαστε στην διάθεσή σας και όλοι είμαστε έτοιμοι να συντονίσουμε τις προσπάθειες των χωρών μελών. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε. Ευχαριστώ. Thank you Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Επίτροπε, που ήρθατε